So, ladies and gentlemen, Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ, θα ήθελα να συνεχίσουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και να σας παρακαλέσω να λάβετε θέσεις. Περνάμε στο σημείο 8 της ημέρησης διάταξης. Ε, είναι ψηφοφορία επί τη σύσταση προς την ύπατη εκπρόσωπο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόταση τη ΥΠΑΤΗ εκπροσώπου τη Ένωση για θέματα εξωτερική Πολιτική και πολιτική ασφαλείας με την υποστήριξη τη Επιτροπή προ το Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση απόφαση του Συμβουλίου και τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη. Η συγκήτρια είναι η κυρία Χίλτε Φάουτμαν. Θέλει το λόγο μήπω όχι. Οπότε πάμε κατευθείαν στη ψηφοφορία. <coughs> Ξεκινάμε με την τροπολογία 65. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α, λάθος, συγγνώμη. Απορρίπτεται. Αυτό πραγματικά θα γράφαμε ιστορία αν ίσχυε. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 69 έχει αποσύρθει. Συμβαστική τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 74. Το κύριο Σαφοζέρ. Υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 73. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 75. Υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 76. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Κάτι λέει ο κύριος Στάνοκ εκτός μικροφώνου όμως. No, this is not... We will I think we can deal with Mr. Uh, individually. Θα το δούμε αυτό διμερώς με τον κύριο Σαφόζερ. 77. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 78 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για την τροπολογία 78. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην 81. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 82 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 84 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 85 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 85. Άρχεται ψηφοφορία. Ένας υπεράριθμος σοσιαλιστής ψηφίζει. Απορρίπτεται με 29 ψήφους υπέρ και 30 κατά. 86. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 87 υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 88 υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 89 υπέρ, κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 89. Άρχεται ψηφοφορία. Closed. Suspended. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα πρέπει να ελέγξουμε και την 90. Άρχεται ψηφοφορία. 90,2. And it's Τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται και αυτή. Ακόμη και υπέρ να δεν αρκεί για να ανατρέψει το αποτέλεσμα. Πάμε στην 91. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 96 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 99 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 99 άρχιτη ψηφοφορία κατά εγκρίνεται 100 υπέρ κατά αποχές μάλλον εγκρίνεται 101 υπέρ κατά αποχές θα πρέπει να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά άρχιτη ψηφοφορία για την 101. Close. Τέλος. Α, απορρίπτεται ή κάποιος λείπει. Ισοπαλή, αλλά απορρίπτεται. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για την 102. Μάλλον ήδη ίδιο αποτέλεσμα θα έχουμε, ισοπαλία δηλαδή. Όχι, όχι, με διαφορά απορρίπτεται. 103 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 104 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 105 έχει αποσυρθεί. 106 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 107 υπέρ, κατά. Αποχές και αυτή απορρίπτεται. 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ κατά αποχές Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 109 του κ. Μεζερίτς άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας και εγκρίθηκε. 110 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 111 καταπίπτει. 112 το ίδιο, 113 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 114 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο, μάλιστα, για την 114 άρχιτη ψηφοφορία. Clearly adopted με διαφορά εγκρίνεται. 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 119 άρχη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 120 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο. Καλώς. Άρχεται η ψηφοφορία για την 120. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Οι φιλελεύθεροι θα πρέπει να σηκώνουν τα χέρια τους για να φαίνεται. 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 124 δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 126 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 126 του κυρίου Νταουνζό. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 127 υπέρ, κατά αποχές. Θα πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά και την 127 του κυρίου Πέτερλε. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος εγκρίνεται. 128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 129 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος και για την 129 άρχιτη ψηφοφορία τέλος εγκρίνεται 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 133 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 133 άρχη ψηφοφορία. Close. It's been adopted. Τέλος, εγκρίνεται. 134, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις. 8, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 9, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. in 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 16 άρχεται η ψηφοφορία It's closed. Τέλος εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ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 31 του κυρίου Μπενιφέ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 34 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος και για την 36 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος απορρίπτεται. 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ κατά αποχές Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 38, κατά την γνώμη μάλλον απορρίφθηκε. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος, απορρίφθηκε όντως. 39 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος και για την 39, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος, εγκρίνεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 40 άρχεται η ψηφοφορία είναι τον Βαλέρο και λοιπόν τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται α όχι λάθος τι γίνεται Τσάρλς περιμένεις την κάρτα ψηφοφορία σου Απορρίπτεται. Με ισοπαλία 30 όλα. Ο Τσάρλς Τάνοκ ε, δεν έχει κάρτα. Πού είναι η κάρτα, στο Λονδίνο? Σαράντα δύο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά το πρώτο τμήμα, αρχή ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας, με διαφορά εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τη 46 την υπερψηφίσαμε, όχι. 48 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 49 άρχιτη ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 52 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 53, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος, απορρίπτεται. 54 υπέρ, κατά αποχές. Απορρίπτεται. 55 υπέρ, κατά αποχές. Απορρίπτεται. 56 υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται. 57 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία υπαριθμών 1. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχεται ψηφοφορία. It's closed. Τέλος, σαφώς απορρίπτεται. 58. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 59. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ κατά αποχές Πολλές τροπολογίες του Φροντζουλίκα. Α την ελέγξουμε ηλεκτρονικά, όμω άρχεται η ψηφοφορία για την 63. Α, τώρα πολύ άσχολος. Τέλος ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά όμως. Τροπολογία 64, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Πάμε στις αιτιολογικές αναφορές. Υπαριθμόν 1. Τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Καταπίπτει. 4. Υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε και τις τροπολογίες 6 και 7 που είναι πανομοιότυπες. Για την αιτιολογική αναφορά 12. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνονται. Και ψηφίζουμε το σύνολο της έκθεσης όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος και εγκρίνεται με 52 ψήφους υπέρ και 7 κατά. Κυρία Λέζινγκ, εκ μέρους ομάδας μου έχουμε συντάξει ε, έκθεση μια ψηφία. Την έχουμε ήδη αποστείλει στη γραμματεία. Ευχαριστούμε. για αυτή την πληροφορία. Υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις. Όχι, επομένως προχωρούμε στο σημείο 9 της μερίσιας διάταξης σύσταση προς Συμβούλιο, Επιτροπή και είπατε εκπρόσωπο της Ένωσης για τη νέα συνολική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουσμπεκιστάν. Μπορούμε να περάσουμε, αν δεν απατώμε ευθύς αμέσω στην ψηφοφορία. Συμβιβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 43 ψήφι υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε τη 43 άρχεται ψηφοφορία. It's closed. This has been rejected. Απορρίπτεται. Τροπολογία 50 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται και αυτή. Συμβιβαστική 8 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβεβαστική 12 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προχωρούμε στην τροπολογία 86 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 87 ψήφι υπέρ κατά αποχές Καλύτερα να ελέγξουμε την 87 του κυρίου Σόλτς. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία, απορρίφθηκε. Συμβιβαστική 13, ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολέγω 89 ψήφι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 90 ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 94 και 95 ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική 14 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 99 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 100 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 101 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 15 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολή 117 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16 ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17 ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολή 128 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται. 134 ψήφι υπέρ, κατά αποχές θα ελέγξουμε την τροπολογία 134, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Συμβιβαστική 19 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 142 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Θεολογικές σκέψεις, ρισάιτας. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θεολογικές αναφορές ετέσνος. Πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές Ελέγχουμε τη δεύτερη τελική αναφορά, το citation 2, την τροπολογία 2 δηλαδή. Πέρας, εγκρίνεται, τρία υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο του σχεδίου σύστασης όπως τροποποιήθηκε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 60 ψήφι υπέρ, 2 κατά. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και περνάμε στο σημείο 10, που είναι η σύσταση προς Συμβούλιο Κομισιών και είπατε πρόσωπο για την ε, θεσμική συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωση ε, και Δυτική Συνομοσπονδίας. εισηγητής ο συνάδελφό μα Φρουντζούλικα. Δεν ξέρω αν θέλει το λόγο. Όχι, δεν τον επιθυμεί. Επομένως, μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Συμβιβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 2 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. ΥΜΚΟ παράγραφος 1. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Είναι τα 2. Υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Ήμκο παράγραφος 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ήντε 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ίντε 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Είναι τα 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ήμκο παράγραφος 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ήμκο παράγραφος 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ήμκο παράγραφος 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τσεκ. Έλεγχο Έλεγχος για την συμβαστική 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία, Εγκρίθηκε. Ήμκο παράγραφος 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 7 συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ίντα 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Απορρίπτεται, συγγνώμη. Ήμκο 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ίντα 5 δεν ψηφίζεται. Ούτε η 6 ούτε η 11 και η Ήμκο 9 ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές δεκτή. 10 Ήμκο υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ήμκο 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ήμτα 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δεν ψηφίζουμε την τα 10. Συμβιβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τοπολογία 65 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11 συμβαστική υπέρ κατά αποχές δεκτή. 70 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 71 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 72 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 73 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 9 διορθώνει ο πρόεδρος. 15 συμβαστική υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ήμκο αιτιολογική α υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 13 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 14 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 15 αποσύρθηκε. 16 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 17 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 16 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 20 τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 21 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 22 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 23 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 24 αποσύρθηκε, 25 υπέρ, κατά, αποχές. Έλεγχος για την 25, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας, εγκρίθηκε. 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 23 υπέρ 33 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές δεκτή. 34 υπέρ κατά Αποχές δεκτή. Αιτιολογικές, αιτιολογικές αναφορές. Αιτιολογική 1. 4 της ΣΥΜΚΟ υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ήμκο 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ήμκο 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ήμκο 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ήμκο 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ήμκο 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Όχι, πίπτη διορθώνει ο πρόεδρος. Ήμκο 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο του σχέδιου έκθεσης άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε. 48 υπέρ, 8 κατά. Πάμε στην επόμενη και τελευταία ψηφοφορία για σήμερα, την έκθεση σχετικά με την έκθεση Επιτροπής για το 2018 για την Τουρκία. Η συγκεκριά μας η κυρία Κατυπήρη. Θέλει πω το λόγο. Όχι, πάμε κατευθείαν τότε στις ψηφοφορίες. Συμβαστική τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Α, έχουμε και μια καλή είδηση. Έχει έρθει η κάρτα του κύριου Τάνοκ. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 56 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, Μάλλον απορρίπτεται, αλλά θα ελέγξουμε καλού κακού. Άρχεται η ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα της 56. Τέλος. Ε, με σαφή διαφορά απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, απόχες. Θα ελέγξουμε και το δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος εγκρίνεται η 57 καταπίπτει πάμε στη συμβαστική τροπολογία 4 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 63 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα έρχεται η ψηφοφορία Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 103 του κύριο Μπέλντερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ναι 106 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 108. Καλώς. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Κατά κράτος.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 157. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 159. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 163. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά τη συμβαστική τροπολογία 13. Τέλος. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 180. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 181 και 182 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτονται. 183 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 184 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 185 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 185 έρχεται η ψηφοφορία. It's closed. Τέλος. Rejected. Απορρίπτεται. 186. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 187 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 188 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 220 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 220. Θέλετε έλεγχο για 220. Καλώς. Άρχεται η ψηφοφορία. Αν και είναι αργά πια. Μας λείπουν 7 ψήφοι. 220 ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος ψηφοφορίας. 62 προς 1. ...221 τώρα, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 18 που είναι, εδώ είμαστε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβεστική 19, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβεστική τροπολογία 20, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 319. Τροπολογία 319. Αγαπητοί φιλελεύθεροι, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 21. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ, κατά, αποχές, Μάλλον απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 13. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τροπολογία 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε στην τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία της έκθεσης, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται 47 προς 7. Διάφορα δεν έχουμε. Η επόμενη μας συνεδρίαση θα γίνει στις 4 Μαρτίου από τις 3 και θα ήθελα να ζητήσω από τα μέλη του Διευρυμένου Προεδρείου να παραμείνουν στην αίθουσα. Θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση του Διευρυμένου Προεδρείου αμέσως.